τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης καθώς και τα εγκεκριμένα κείμενα ε, διατίθενται. Έχετε διαφωνίες, αντιρρήσεις, όχι. Οπότε και θεωρώ.